Ladies and gentlemen, dear colleagues, good morning. As uh, you can imagine, I'm replacing our chair. Οπότε καταλαβαίνετε, ανεκαθιστώ τον κύριο Ρόλ, τον πρόεδρό μας, που είναι συνεδρίαση του ΕΛΚ στο Παλέρμο. Χαίρομαι όμως που βλέπω ότι ορισμένοι του ΕΛΚ έχουν μείνει εδώ. Ε, η συζήτηση στην Επιτροπή μας ε, θα ακολουθήσει. Θεωρώ ότι έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη και καθότι δεν έχω να κάνω ανακοινώσεις, ε, προτείνω να ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση για την έκθεση Jordan Sitchell για την διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Σήμερα θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή έχει, έχει γίνει μια ε, πρώτη ε, ανταλλαγή απόψεων. Η, η προθεσμία για την ε, κατάθεση τροπολογιών ήταν 12 Απριλίου και θα παρακαλούσα την Ρωμάνα να μας παρουσιάσει την κατάσταση όσον αφορά τις τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέρφους που έχουν υποβάλει διάφορες τροπολογίες. 293 τροπολογίες έχουμε λάβει, πράγμα που δείχνει ότι είναι πολύ σημαντική, ότι θεωρείτε εσείς πολύ σημαντική την έκθεση αυτή. Η οδηγία που συζητάμε είναι επίσης πολύ σημαντική και είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το κείμενο μαζί. Ε, προσπάθησα να ομαδοποιήσω τις ε, τροπολογίες όσον αφορά το περιεχόμενό τους ε, και θα σας κάνω τώρα μια σύντομη παρουσίαση και θα σας ε, πω και τη δική μου γνώμη για αυτές. Πρώτον, θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν τροπολογίες που αναφέρουν την καταστροφή στη Ιαπωνία, τα γεγονότα στην Φουκουσίμα. Πιστεύω ότι πράγματι μπορούμε να εξοπλίσουμε τα γεγονότα αυτά ως σημείο αναφοράς για να τονίσουμε την ε, σημασία των επαρκών ε, προτύπων ασφαλείας ε, για τα ραδιενεργά απόβλητα και τα αναλωμένα καύσιμα. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε συμβιβασμό στο θέμα αυτό. Ωστόσο, δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει για το λόγο αυτό να απορρίψουμε την οδηγία. Ακριβώς εξαιτία των όσων συνέβησαν στην Φουκουσίμα είναι τόσο πιο σημαντική η οδηγία αυτή. Υπάρχουν και πολλές ε, τροπολογίες που λένε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την πυρηνική ενέργεια, αλλά αυτό πιστεύω ότι δεν εμπίπτει στην εντολή μας, δεν εναπόκειται σε εμάς να το αποφασίσουμε αυτό, γι' αυτό τις απορρίπτω. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες σχετικά με την τροποποίηση της νομικής βάσης. Να αναφερόμαστε δηλαδή στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν θα εκφράσω θέση για το θέμα αυτό σήμερα, διότι περιμένω την γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ήδη Έχουμε ε, υποβάλει σχετική ερώτηση στην Επιτροπή αυτή. Η επόμενη ομάδα τροπολογιών έχει να κάνει με οικονομικούς πόρους. Εγώ η ίδια έχω τροποποιήσει το κείμενο, ωστόσο λάβαμε και άλλες τροπολογίες ε, για να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, να υπάρχουν ε, έλεγχοι και αντίβαρα και υπάρχουν και τροπολογίες σχετικά με την αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και εδώ σε συμβαστική τροπολογία. Μάλλον θα πρέπει να έχουμε δύο συμβαστικές τροπολογίες, μία για τα εκτιμώντας και μία για το διατακτικό του κειμένου. Περίπου 15 ή 20 τροπολογίες σχετίζονται με την ε, ορολογία. Κάποιοι θέλουν να μιλάμε για τελική αποθήκευση, άλλοι θέλουν για, να μιλάμε για τελική διάθεση. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την, ε, τους όρους που ήδη έχουν γίνει αποδεκτοί, οι οποίοι ε, κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στην αποθήκευση που δεν είναι μόνιμη λύση και τη διάθεση που αποτελεί μόνιμη λύση. Μιλάμε λοιπόν για τελική διάθεση με τη δυνατότητα αναστρεψιμότητας. Ελπίζω ότι σε συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στην χρήση αυτών των όρων. Αυτό πιστεύω ότι θα κάνει πιο ε, καθαρό το κείμενό μας. Ε, μπορώ όμως ε, να δεχτώ τον όρο τελική αποθήκευση αντί για τελική διάθεση, διότι η τελική αποθήκευση δεν σημαίνει ότι μιλάμε για κάποια οριστική λύση. Επίσης μιλάμε για την βαθιά γεωλογική διάθεση ε, ε, ελπίζω θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες λένε ότι αυτή είναι μία επιτεύξιμη λύση και ε, βιώσιμη λύση. Ωστόσο πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή σε περίπτωση που βρεθούν άλλες λύσεις οι οποίες να τα πρότυπα ασφαλείας. Ελπίζω λοιπόν και εδώ πέρα να καταλήξουμε σε συμβαστική τροπολογία. Επίσης είχαμε κάποιες τροπολογίες σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και εδώ θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστική τροπολογία διότι έχουν υποβληθεί διάφορες τροπολογίες ιδιαίτερα από την Επιτροπή Εργασίας. Επίσης ε, λάβαμε κάποιες τροπολογίες σχετικά με την διασυνοριακή συνεργασία. Πιστεύω ότι είναι καλό να επιτρέψουμε την ε, περιφερειακή και διαπεριφερειακή συνεργασία, διότι έτσι μπορούμε να συγκεντρώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό και τις ε, δεξιότητες των ανθρώπων. Ωστόσο, δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι αυτή ε, η διασυνοριακή διάθεση θα πρέπει να είναι δυνατή παρά μόνο εάν ένα κράτος έχει μικρό όγκο ραδιενεργών αποβλήτων. Τι σημαίνει όμως μικρός όγκος, γι' αυτό εγώ θα απέριπτα την ιδέα αυτή. Ε, υπάρχουν επίσης κάποιες ε, τροπολογίες ε, σχετικά με τις τεχνικές λύσεις. Για παράδειγμα, το πότε θα πρέπει τα αναλωμένα καύσιμα να ε, μεταφέρονται σε ξηρές ε, αποθήκες ραδιενεργών αποβλήτων, πότε θα πρέπει να γίνεται επανεπεξεργασία αυτών των ε, καυσίμων. Αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να τα λύσουν οι πυρογνώμονες, Εμείς όμως ωστόσο πρέπει να θέσουμε τα πολιτικά κριτήρια. Κάποιοι από εσά αναφερθήκατε στις εθνικές αρχές ε, ελεγκτικές αρχές. Ε, υπήρχαν τροπολογίε ε, σχετικά με την σαφή εντολή και τις προτεραιότητες των αρχών αυτών. Πιστεύω όμω ότι εδώ πρέπει να θέσουμε ένα όριο, διότι αυτή είναι μια γενική οδηγία. Δεν είναι εδώ ο χώρο να ορίσουμε ακριβώς τι εντολές των εθνικών αρχών. Επίση, υπήρξαν κάποιες τροπολογίες ε, σχετικά με την ε, βιωσιμότητα και εξετάζω ακόμα εάν ε, αυτές συνάδουν με την σύμβαση του Παρισιού. Όπως ήδη έχω πει, δεν πρόκειται για οδηγία όπου ψηφίζουμε υπέρ ή κατά της ατομικής ενέργειας, ούτε έχει να κάνει με την βαθμιαία κατάργηση και αντικατάσταση της σε, με άλλες πηγές. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είναι εδώ κατάλληλος χώρος να λύσουμε τα θέματα αυτά. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει 100% ασφάλεια ούτε στον χώρο της ε, πυρηνικής ενέργειας ούτε ε, όσον αφορά άλλες μορφές ενέργειας. Γι' αυτό απορρίπτω όλες τις τροπολογίες που μιλούν για ασφάλεια 100% διότι είναι μη ρεαλιστικές. Στηρίζω τις τροπολογίες που αναφέρονται στο υψηλότερο, πιθανό, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας. Ε, αυτές τις ε, τροπολογίες φυσικά θα τις στηρίξω. Την ε, προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την ρήτρα αποσύρση το sunset close που πρότεινε η Φιώνα Χολ, που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα. Βρίσκω κάπως ασθενή αυτή την τροπολογία. Μετά από 15 χρόνια προτείνει εκείνη ε, προθεσμία. Πιστεύω όμως ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το λύσουμε σε συνάντηση με τους κοιόδης συζητητέ. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για όλες τις τροπολογίες που υποβάλλατε και θα ακούσω προσεκτικά όλες σας τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόδο. Η συζήτηση αρχίζει τώρα επί του θέματο. Καταρχήν θα ακούσουμε τους κοιόδης συζητητέ. Η κυρία Ρεμπέκα Χάρψ είναι νομίζω η πρώτη που ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν αναφερθώ στην, στο σχέδιο χρηματοδότησης και στις απολογές που έχουν υποβληθεί, θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που είχα πει και στην τελευταία συνάντηση των σκιωδών εισηγητών. Θυμόσαστε σίγουρα μια που είσαστε ενεργά μέλη της Επιτροπής αυτής, θα θυμόσαστε λέω τη συζήτηση που είχαμε για την οδηγία, για τα πρότυπα ασφαλείας, για τους πυρηνικούς σταθμούς Ενέργεια. Μια οδηγία που είναι ήδη δύο ετών και που λίγες μέρες μετά τη Φουκουσίμα όταν αρχίσαμε να συζητάμε με τον Επίτροπο για τα στρέστες είδαμε ότι είχαμε κάνει ένα τεράστιο λάθος όταν υιοθετήσαμε αυτήν την οδηγία γιατί η οδηγία δεν προβλέπει φιλόδοξα δεσμευτικά πρότυπα ασφαλείας. Το πρόβλημα στη διατύπωση των κοινών στρέτες είναι ότι μια που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινά ε, πρότυπα ασφαλείας αυστηρά, δεν μπορεί να κλείσει αυτό το κενό τώρα. Και γι' αυτό ε, θα πρέπει να συζητήσουμε για άλλη μια φορά το θέμα των φιλοδόξων προτύπων ασφαλείας για την πυρηνική ενέργεια και φοβούμε ότι το ίδιο σφάλμα που κάναμε όταν ε, ορίσαμε ε, την οδηγία για τα μέτρα αυτή ασφαλείας κάνουμε το ίδιο λάθος λέω όταν καθορίζουμε τα πρότυπα για την τελική απόθεση και την διαχείριση των αποβλήτων. Ακριβώς η έκθεση της συζητήτρες της Επιτροπής αποδυναμώνει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. η δήλωση ότι ορίζουμε υψηλού επίπεδου δεσμευτικά πρότυπα δεν ε, αποδεικνύεται με την έκθεση αυτή. Και θα ήθελα πραγματικά να ξανασυζητήσω εάν αυτό είναι η πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη Φουκουσίμα. Δηλαδή να υπάρχει πάλι μία πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήδη δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη όσον αφορά τα πρότυπα ασφαλείας και τις διαδικασίες για τις τοποθεσίες τελικής απόθεσης να αποδυναμώνεται επιπλέον με τη δική μας έκθεση. Έτσι αξιολογώ εγώ αυτό που υπάρχει τώρα επιτάπητος και για το οποίο διαφαίνεται μια πλειοψηφία στην Επιτροπή. Θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά γιατί η δημόσια συζήτηση νομίζω μετά την Φουκουσίμα η απόσταση η χρονική δεν είναι τεράστια, η κατάσταση δεν είναι υποέλεγχο. Ιδίως υπήρχαν και κάποιοι τις δεξαμενές αναπόθεσης ε, που δεν ήταν καλά ασφαλισμένη, Αυτό αυξάνει το πρόβλημα, το δυστύχημα της Φουκουσίμα και γι' αυτό θα ήταν καλό τα τελικά ε, αποτελέσματα είναι πιο αυστηρά από ό,τι επιθυμούν ορισμένοι συνάδελφοι. Ένα αυτό. Ένα άλλο που θα ήθελα να αναφέρω. Είναι δύο σημεία τα οποία έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό που υποβάλλαν οι σκιώδησηγητές γιατί θεωρώ ότι ακριβώς μετά την δήλωση του ε, Επιτρόπου Ενεργείας θα αναγκαστούμε να κριθούμε πάνω σε αυτά. Το πρώτο σημείο αφορά το μέλλον των εξαγωγών των αποβλήτων από πυρηνικές εγκαταστάσεις είπε ο Επίτροπος ξεκάθαρα ότι θέλει να αποκλείσει στο μέλλον να εξάγονται τα απόβλητα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπε τόσο συχνά όσο δεν το είχε ποτέ κανένας υψηλά ιστάμενος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι απάντησε και σε ένα πρόβλημα. Δηλαδή μέχρι στιγμής η κατάσταση ήταν οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες να γίνονται ασίδωτα. Γιατί σε τρίτες χώρες δεν έχουμε τη δυνατότητα της ε, απόθεσης των αποβλήτων αυτών σύμφωνα με τις δικές μας ιδέες ασφαλείας. Και από αυτού θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν σήμερα πώς τοποθετείται στη δική της πρόταση σήμερα η Κομισιόν. Εξακολουθεί δηλαδή να πιστεύει ότι αυτό που είπε ο Επίτροπος και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το δηλώνει, είναι σημαντικό, δηλαδή να απαγορευτούν οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Επίσης θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει και θα ήταν χρήσιμο αυτό για τη συζήτηση με την εισηγήτρια, ποιες είναι εκείνες οι χώρες στις οποίες θα μπορούσαμε να φανταστούμε να εξάγουμε ε, τα απόβλητα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες χώρες και πού ακριβώς τις χώρες αυτές θα εξαγάγαμε αυτά τα απόβλητα και κατά πόσον τότε θα ακολουθήσουμε την οδηγία 117 Ευρατόμ του 2006 του Συμβουλίου ή υπάρχουν και συζητήσεις να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Και θα ήθελα επίσης να ακούσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση με το Συμβούλιο πώς ε, θεματοποιεί τον στόχο της απαγόρευσης των αποβλήτων, το, της εξαγωγής των αποβλήτων γιατί σας είπα, το είπε πλειστάκης ο Επίτροπος κύριος Ότιγκερ ότι θα απαγορευτούν αυτές οι εξαγωγές δηλαδή. Αλλά οι φήμες που ακούγονται και διαδίδονται στις Βρυξέλλες δεν είναι πολύ καλές. Και ιδίω στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Φουκουσίμα. Αυτό που θα ήθελα επίσης να μου πει η Κομισιόν και που συζητήθηκε στη τελευταία συνάντηση των σκιωδών εισηγητών με την εισηγήτρια το πώς ε, διαβλέπει η Κομισιόν α, τις ε, προτάσεις της εισηγήτριας για την λεγόμενη safety case. Η Κομισιόν το είχε συγκεντρώσει το θέμα αυτό σε μία παράγραφο της οδηγίας. Η εισηγήτρια θεώρησε ότι θα ήταν καλό να το με αυτό παντού, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ιδέες για αιτιολογικές σκέψεις, για το safety case να υπάρχουν εδώ και εκεί. Αυτό εμένα με ενοχλεί, δεν μου φαίνεται πολύ καλό, γιατί μου φαίνεται ότι αυτό επιπλέον αποδυναμώνει την πρόταση της Κομισιόν. Τέλος, για τη σημερινή συζήτηση θα ήθελα να αναφερθώ στον ισχυρισμό της εισηγήτριας ότι ο στόχος δεν είναι να επιτύχουμε υψίστη ασφάλεια. Ε, εγώ καλύτερα από πολλούς ξέρω, γιατί ασχολούμαι εδώ και 30 χρόνια με το θέμα της ελληνικής αναπόθεσης, ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να επιτευχθεί 100% ασφάλεια. Όμως ως πολιτική θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε την ε, υψηλότερη δυνητή ασφάλεια. 50 χρόνια μετά τη σε υπηρεσία του πρώτου πυρηνικού αντιδραστήρια έχουμε 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στερεά απόβλητα που δεν ξέρουμε να τα κάνουμε. Από εκεί διαφαίνεται το πόσο δύσκολο είναι να επιληθεί αυτό το θέμα των ε, πυρηνικών αποβλήτων. Και αν δεν υπάρχει λύση, αυτό είναι ένα εμπόδιο για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Γιατί θα ήθελα να ακούσω, ιδίω μετά τις εμπειρίες της Φουκουσίμα, τις χώρες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σεισμών, πώς μπορούν να υπάρχουν βαθιά ε, γεωλογικά ε, τοποθεσίες τελικής εναπόθεσης. θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτού του τύπου τις προτάσεις μέσα στα πλαίσια της πρότασης ηγήτριας. 100% δεν θα υπάρχει ποτέ, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Και η έκθεση απέχει πολύ αυτό, γιατί ούτε ο σεισμός σαν κίνδυνο δεν αναφέρεται, ακόμα και μετά τη Βουκουσίμα. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mrs. I'd like uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Κινινόφσκι από το ECR να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ε, καταρχήν θα ήθελα ε, να επενέσω την ε, δουλειά της ε, εισηγήτριας. Ε, είχαμε τα γεγονότα στην Ιαπωνία, τα οποία έχουν περιπλέξει πολύ την συζήτηση και πιστεύω ότι είναι θετική η προσπάθεια στη... έκθεση αυτή να κρατήσουμε μια ορθολογιστική στάση στην έκθεση αυτή δεν ε, μπορούμε να ασχοληθούμε με το συνολικό πρόβλημα της ε, ενεργειακής πολιτικής. Εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα. Η εμπειρία της ε, Φουκουσίμα μας δίνει τη δυνατότητα να τονίσουμε τα σημαντικά και να συμπεριλάβουμε τις πληροφορίες που είναι σημαντικές για το κοινό. Είναι σημαντικό να γίνεται κατανοητό ότι μιλάμε για επικίνδυνα απόβλητα, από την άλλη όμως ε, να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν να λύσουν τα θέματα αυτά. Επίσης θα πρέπει να έχουμε αυστηρούς κανόνες και πρότυπα για την ε, διαχείριση των ε, επικίνδυνων ουσιών. Η πολιτική μας ομάδα θα ήθελε όσον αφορά την ε, αποθήκευση ε, βαθιά μέσα στη γη ε, να τονιστεί το θέμα αυτό, διότι δεν ξέρουμε κατά πόσο θα εξελιχθεί γρήγορα η τεχνολογία και μπορεί να είναι πολύ ακριβή η εξέβρεση λύσης για την οριστική διάθεση των αποβλήτων. Ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ε, τεχνικά εφικτές λύσεις και θα πρέπει να φροντίσουμε οι χώροι αποθήκευσης ε, να παραμένουν υπό έλεγχο. Επίσης θα στηρίξουμε τις προσπάθειες ε, για κοινέ διαπεριφερειακές λύσεις, ε, διότι η συνεργασία, ε, η ευρύτερη συνεργασία σίγουρα είναι σημαντική και όσον αφορά τις πτυχές ασφαλείας. Ε, θα πρέπει να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις υπό τις ε, υπάρχουσες προϋποθέσεις. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε να μας ε, παρασύρουν τα τραγικά γεγονότα της Φουκοσίμα. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτά. Έχουν γίνει τεχνικά λάθη στην Φουκουσίμα και θα πρέπει να εξάγουμε από αυτό συμπεράσματα. Το βασικό πρόβλημα δεν ε, ήταν ο σεισμός, ε, αλλά το κύμα τσουνάμι. Είναι πολύ σημαντική η σωστή πληροφόρηση των πολιτών. Θα πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι εδώ μιλάμε για επικίνδυνα ραδιενεργά απόβλητα και ότι είναι απαραίτητο να βρούμε τεχνολογικές λύσεις σε υψηλό επίπεδο. Η πολιτική μας ομάδα θα στηρίξει την εξέβρεση καλύτερων λύσεων για την διαχείριση αναλωμένων καυσίμων. Συμφωνώ με την κυρία Χάρμς ότι η συζήτηση δεν θα είναι εύκολη. Θα πρέπει όμως να επικεντρωθούμε στην ε, σωστή πληροφόρηση και τη βελτίωση των ε, κανόνων για την ε, διάθεση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Ήδη υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Και ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε και μια άλλη πτυχή, το σε ποιες χώρες μπορούμε να εξάγουμε τις σχετικές τεχνολογίες. Δεν μιλώ για την ε, εξαγωγή ραδιενεργών αποβλήτων ε, απαραίτητα, αλλά Ίσως είναι και αυτό ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να διατίθενται τα ραδιενεργά απόβλητα με τρόπο ώστε να μην μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κατάξυσης από τρομοκρατικές οργανώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε ορθολογιστικέ λύσει ώστε να βελτιώσουμε τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και διανεργών αποβλήτων. Ευχαριστώ. S&D. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω με μια ευχή σε ό,τι αφορά την ε, ημερησία διαταξή μας, την ατζέντα μας. Ε, στην δεύτερη ολομέλεια των σε συζητείται αυτό το θέμα, μετά το Συμβούλιο δηλαδή. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικό αν η Επιτροπή καταβάλει κάποιες προσπάθειε έτσι ώστε η δική μα γνωμοδότηση να φτάσει στο Συμβούλιο πριν να λάβουν τελική απόφαση και θετήσουν την νομοθεσία. Γιατί ε, αυτό ανήκει στην διακυβερνητική διαδικασία υπό την Ευρατόμ, τη συνθήκη τη Ευρατόμ. Και αν ε, κατορθώσουμε εμεί να έχουμε έτοιμη την γνωμοδότησή μα εν τον χρόνο, μπορεί να κατορθώσουμε να βρούμε μια λύση, να επιταχύνουμε τη διαδικασία κατά δύο εβδομάδες. Ε, θα μπορούσαν ε, να τη διαβάσουν την έκθεση οι βουλευτέ και να δούμε πόσοι ψηφίζουν και προς ποια κατεύθυνση για το θέμα. Ελπίζω να βρούμε εδώ μία λύση και αν είναι δυνατόν να επιταχύνουμε θα ήταν κάτι θετικό. Φυσικά, για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι ότι θέλουμε να επιδιώξουμε την ε, πλειοψηφία μεταξύ των πολιτικών ομάδων όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε, γιατί έτσι θα αποδείξουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι σοβαρός εταίρος και κινείται προς μια κατεύθυνση. Βλέπω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσει ότι, και, συμφωνεί ότι πρέπει να αναλυφθεί δράση και εφόσον όλοι αναφέρουν το Φουκοσιμία και εγώ πρέπει να την αναφέρω. Αν ε, υπάρξει διεθνές πρότυπο και μια διεθνής διαδικασία για το τι θα κάνουμε με τα πόβλητα τότε ε, ίσως ε, θα περιοριστούν τα θέματα που αντιμετωπίζουμε. εκεί έτσι λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι όσα γίνονται σήμερα παγκοσμίω δεν αρκούν και πρέπει να αναλυφθεί δράση. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο έχει περιορισμένο ρόλο, λόγω της συνθήκης Ευρατόμ, αλλά και επειδή όλα τα θέματα που συνδέονται με το ενεργειακό μείγμα ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν, αν σε αυτές τις τροπολογίες που είναι υπό την ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, καλό θα ήταν να έχουμε μια γνωμοδότηση από, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ομάδα των σοσιαλιστών δεν θα είναι ενωμένη. Ω και ηγήτρια, εγώ δεν είμαι έτοιμη να πω ποια θα είναι η τελική άποψη τη ομάδα μου, γιατί μάλλον θα έχουμε μία ε, λύση πολύχρωμη, αν μπορώ να την πω έτσι. Θα πρέπει να Έχουμε, ε, εγώ προσπάθησα να οθήσω και να υπάρξει συμβιβασμό μέσα στην ομάδα. Έχω τέτοια ευθύνη ω και Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε αποκλίνουσες απόψεις σε πάρα πολλά θέματα και οι συνάδελφοι που είναι και εδώ, που παρευρίσκονται εδώ, θα εξηγήσουν τη δική τους άποψη. Αλλά σίγουρα σε ορισμένα πράγματα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και ευαισθησία του κοινού, γιατί μόνο με την κοινή γνώμη μπορούμε να κερδίσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να γνωστοποιήσουμε το ζήτημα αυτό. Δεύτερον, πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό στις τροπολογίες και ε, φυσικά η ύψιστη προτεραιότητα για μας πρέπει να είναι το εργατικό δυναμικό. Οι άνθρωποι που εργάζονται με τέτοιες επικίνδυνες ουσίες ε, πρέπει να προφυλάσσονται και επίσης πρέπει να ε, παρέχονται και με ακροπρόθεσμα πρότυπα ε, επιστημονικά και πρότυπα ποιότητας. Ε, το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης είναι πάρα πολύ χρήσιμο Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε πολύ σοβαρά εκείνες τις τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές στην Επιτροπή Απασχόλησης. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε την πόρτα για πιθανή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη, αλλά φυσικά αν οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, ουσιαστικά οικοδομούν ε, ε, ένα σημείο απόθεση των αποβλήτων και το ίδιο κάνει και η Ρωσία. Εμεί πιθανότητα θα έχουμε 27 χώρες που θα έχουν διαφορετικά συστήματα για την τελική διάθεση των αποβλήτων. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Εδώ μιλάμε για σχεδιασμό για χιλιάδες χρόνια στο μέλλον και νομίζω ότι συμφωνούν οι συνάδελφοι ότι πολύ συχνά έχουν αλλάξει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης τα τελευταία 100 χρόνια. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι σε χίλια χρόνια μπορεί και να έχουν αλλάξει τα σημερινά σύνορα των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε τις καλύτερες λύσεις και όχι βάση πολιτικών σύνορων και πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα για πιθανή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Πιστεύω ότι το ζωτικό θέμα, το κριτικό σημείο είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Θα πρέπει να έχουμε και τους χρηματοδοτικούς πόρους που θα πρέπει να εξασφαλιστούν και να εξοικονομηθούν ε, παρά την κρίση. Γιατί είδαμε ε, πόσο ε, εύκολα χάνονται οι πόροι στο χρηματιστήριο παραδείγματο χάρη. Έτσι λοιπόν είναι επιτακτικό να εξεύρουμε μία λύση έτσι ώστε οι χρηματοδοτικοί πόροι να μην λείπουν όταν χρειάζονται. Να μην λείπει η χρηματοδότηση, αλλά δεν μιλάμε μόνο για τη συλλογή, αλλά και για τη χρήση των πόρων αυτών. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που πρέπει να συζητήσουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις που θα καθοριστούν και τι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι την ευθύνη πρέπει να την έχει η βιομηχανία, ο τομέας. Συζητήσαμε πολύ αυτό το θέμα, πώς πληρώνει ο Ριπένον. Συζητήσαμε την αρχή αυτή για αν τα ισότοπα παράγονται σε μια χώρα και εξάγονται σε ποσοστό 60% σε άλλη χώρα, τότε ποιο ε, είναι ο Ριπένον, αυτός ε, που παρήγαγε ή αυτός που χρησιμοποίησε τα ισότοπα. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και να δούμε τι ακριβώ σημαίνει, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να πιέσουμε τη βιομηχανία τελικά να αναλάβει την τελική ευθύνη. Δεν είναι υποχρέωση του φορολογούμενου να πληρώσει. Και πιστεύω ότι ως σοσιαλιστές θα συμφωνήσουμε από αυτού. Εξακολουθούμε να έχουμε και πάλι κάποια προβλήματα με τις τροπολογίες με τον ορισμό των αποβλήτων. Τα κράτη-μέλη έχουν αποκλίνοντες ορισμούς. Ορισμένα κράτη-μέλη διαιρούν ε, τα πόβλητα σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί ορισμοί σε διάφορες χώρες. Πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω από αυτό και έχουμε και την τελική και την έσχατη διάθεση και την ε, προσωρινή ενδιάμεση διάθεση. Οι ορισμοί δεν είναι εντελώ ξεκάθαροι. Ε, αλλά πρέπει να δούμε και το θέμα της λύσης προσπαθήσουμε να βρούμε μια σειρά. Και να κλείσω με το εξή, συνάδελφοι. Κάτι που πρέπει να υποθεί. Αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι όταν υιοθετήσουμε οποιαδήποτε είδο νομοθεσία και ψηφιστή νομοθεσία, στη συνέχεια υπάρχει και δράση. Υιοθετήσαμε την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια πριν δύο έτη και μόνο τρία κράτη-μέλη την υιοθέτησαν σε εθνικό επίπεδο. Και αυτά τα κράτη-μέλη ασκούν ιδιαίτερη κριτική στην πυρηνική ασφάλεια και ε, υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό μεταξύ των κρατών μελών και όταν συζητείτε, ε, σε πέδο 27 βλέπουμε ότι στη συνέχεια στην εθνική του επικράτεια δεν θέλουν να θετήσουν αυτή την νομοθεσία. Εμείς ε, όταν εκπονούμε την νομοθεσία δεν το κάνουμε για λόγους βιβλιογραφίας για να έχουμε εδώ βιβλιοθήκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά γιατί θέλουμε να εφαρμοστεί. Σας ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν ακόμη δύο σκιώδεις ε, από τους Φιλελευθέρους και από την ΚΟΕ που δεν βλέπω στην αίθουσα. Δεν δώσω το λόγο στους υπολείπους. Ο κύριος Βιδέλ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Χάρμς, Μιλήσατε για 200.000 κυβικά ε, μέτρα. Νομίζω ότι ε, ένα μηδενικό ε, λάθος κάνατε. Διότι αν πολλαπλασιάσουμε επί 40 χρόνια την ετήσια παραγωγή, ε, απλά το λέω, φυσικό είμαι, καταλαβαίνετε, τα μηδενικά έχουν σημασία. Ε, μπορείτε να το ελέγξετε πάντως. Όπως και να έχει, 293 τροπολογίες είναι μεγάλος αριθμός και αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η έκθεση του Κοινοβουλίου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Επιτροπής, πράγμα πολύ λογικό. Εάν εξετάσουμε προσεκτικά αυτόν τον μεγάλο αριθμό τροπολογιών, βλέπουμε ότι ουσιαστικά αναφέρονται σε μικρό αριθμό θεμάτων ε, που ε, αντικατοπτρίζουν όμως διαφορετικές ε, ιδεολογικές προοπτικές και αυτό λογικό είναι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές που θεωρώ τις πιο σημαντικές. Καταρχήν βλέπουμε ότι σημαντικός αριθμός τροπολογιών αναφέρεται στους ε, ορισμούς αποθήκευσης και διάθεσης. Αυτοί που υπέβαλαν τροπολογίες θέλουν να αλλάξουν ε, οι ορισμοί αυτοί. Είμαι βέβαιος ότι όλες αυτές οι τροπολογίες θέλουν ε, να αποσαφηνίσουν τους ορισμούς αυτούς. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι πληρούν το στόχο τους, διότι στην πρόταση της Κομισιόν τα πράγματα είναι αρκετά ε, σαφή. Η αποθήκευση είναι προσωρινή, η διάθεση είναι μόνιμη. Οι τροπολογίες αντικατοπτρίζουν το εξή σημαντικό, το να λαμβάνεται υπόψη η, ε, η πιθανή ε, επιστημονική πρόοδος που θα σημειωθεί στο μέλλον. Κυρία Τζόρνταν, το θέμα αυτό μάλλον μπορεί να λυθεί με συμβιβαστική τροπολογία η οποία να αναφέρεται στην αναστρεψιμότητα ή κάτι τέτοιο. Η αποθήκευση όμως και η διάθεση, ε, οι δύο αυτοί ορισμοί είναι απόλυτα σαφείς, οι δύο αυτοί όροι είναι απόλυτα σαφείς όσον ε, αφορά... Αριπόζητορις, ε, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, δεχόμαστε την εξαγωγή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεύτερον, ε, αν το δεχτούμε αυτό, τι γίνεται με την ευθύνη το, του κάθε κράτους μέλους να διαχειρίζεται τα δικά του απόβλητα. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, είναι σαφές ότι η Κομισιόν θέλει να απαγορεύσει την δυνατότητα εξαγωγής αποβλήτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πολλές τροπολογίες δείχνουν ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να εξάγουν εκτός της ε, Ένωσης και γι' αυτό θεωρώ ότι η λύση που παρουσίασαν ε, κάποιοι ε, οι ε, συνάδελφοι θεωρούν ότι το ε, εξάγον κράτος μέλος ε, διατηρεί την ευθύνη. Αυτό θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να είναι και αποτρεπτικό. Και να κάνει τα κάτι μέλη να είναι πιο αυστηρά όσον αφορά την διάθεση τουλάχιστον εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είναι σαφές ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της ε, διαχείρισης ε, των αναλωμένων καυσίμων και των διανεργών αποβλήτων. Θα θυμάστε τη συζήτηση που είχαμε το 2001, ήταν, ε, δεν θυμάμαι, τότε που συζητούσαμε την προηγούμενη οδηγία, η οποία τελικά κόλλησε στο Συμβούλιο. Αλλά να καταλάβουμε το εξής. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υιοθετήσει διαφορετικό τρόπο διασφάλισης ε, των πόρων αυτών όταν χρειαστούν. Εάν όμως θέλουμε να μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες ε, σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει αυτό, τότε θα μπλέξουμε. Γι' αυτό λοιπόν μια οδηγία θέτει κάποιες γενικές αρχές. Μια οδηγία δεν είναι κανονισμός. Θέλουμε γενικές αρχές λοιπόν. Η γενική αρχή θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι οι πόροι όταν έρθει η ώρα να τους χρησιμοποιήσουμε. Εάν όμως μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες, τότε θα συγκρουστούμε με κάποια κρατημέλη και αυτό δεν είναι καθόλου επικοδομητικό. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Βιδάλ Καγουάδρας. Να ζητήσω από την κυρία Βαν Μπρέντ τώρα να πάρει το λόγο και να τη ζητήσω να μας παρουσιάσει ορισμένες υπολογίες που καταθέσαμε μαζί. Γιατί δυστυχώς εγώ θα πρέπει να φύγω νωρίτερα και δεν θα έχω την ευκαιρία να πάρω το λόγο. Μάλιστα θα το κάνω, Άννη. Προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη, αγαπητοί συνάδελφοι γιατί η συζήτηση αυτή είναι ευρύτατη. Έχω υποβάλει μια σειρά τροπολογιών που θα συζητηθούν, αλλά οπωσδήποτε ιδίω οι σκιώδε εισηγητέ έχουν πάρα πολλή εργασία μπροστά του. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν την άποψή μου για την πυρηνική ενέργεια στην οδηγία αυτή δεν συζητάμε όμως κατά πόσο θα εγκαταλείψουμε τη μέθοδο αυτή στην ενέργειας ή όχι. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί αλλού. Εδώ χρειάζομαστε στην Επιτροπή μας μία συνένεση για να πούμε ότι θα πρέπει οι απαιτήσει ασφαλείας να είναι οι υψηλότερες δυνατές. Αυτή είναι η επιθυμία που έχουν όλοι νομίζω. Δεν χρειάζεται να αμφισβητήσουμε, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τη μορφή που θα πάρει κάτι τέτοιο. Αλλά μετά τη Φουκουσίμα νομίζω όλοι ξυπνήσαμε. Βέβαια, δεν χρειαζόταν να φτάσουμε εκεί. Γιατί τα πυρηνικά απόβλητα και η τελική αναπόθεση, τα αναλωμένα καύσιμα κλπ. είναι τόσο πολύπλοκα θέματα και πρόκειται για τεράστιες χρονικές περιόδους, όχι χιλιάδες χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδων. Δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό. Δεν ήταν λοιπόν παράλογο μία χώρα να θέλει να το επιλύσει από μόνη της. Και ε, ε, ε, μετά από 100.000 χρόνια τα σύνορα δεν θα παίζουν κανένα ρόλο είναι σημαντικό να βρει τη λύση η Ευρώπη. Και είναι περίεργο ότι κατασκευάζουμε πάντα τα, τους ποινικούς αυτούς σταθμούς στα σύνορα χωρίς να υπάρχουν κοινωτικές λύσεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Αυτό είναι σημαντικό και σε αυτή τη συζήτηση και σε όλες τις μελλοντικές συζητήσεις. Θα πρέπει πάντα να τονίσουμε ότι είναι δυνατή υψηλή ασφάλεια, υψηλό επίπεδο ασφαλείας μόνο εάν δεν εξάγουμε αυτούς τους πυρηνικούς σταθμούς και να λέμε εντάξει για την ασφάλεια θα πρέπει να ασχοληθούν οι, άλλοι εκείνοι που την αγοράζουν. Όχι. Ο έλεγχος ασφάλειας θα πρέπει να γίνεται από ε, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και ανεξάρτητες ε, ομάδες. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε διαμακρών. Έχω υποβάλει επίσης ε, τροπολογίες για την υγεία των εργαζομένων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδίω για αυτά που είδαμε να διαμείγονται στην Φουκουσίμα. Η καθημερινή ε, εργασία είναι πολύ σημαντική και η μέθοδος που ακολουθείται εκεί θα πρέπει να δούμε πού θα τοποθετήσουμε τους ανθρώπους. Πώς μπορούν ε, να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν, ε, παραλλήλου όμως να σεβόμαστε την υγεία τους. Και κάτι που δεν καταλαβαίνω καθόλου. Είναι περιορισμένο το πεδίο εφαρμογή οδηγία. <coughs> Ίσως για κάποιες πυρηνικές χρήσεις, να μπορούμε να πούμε αυτή είναι καλύτερη, εκείνη δεν είναι τόσο καλή, αλλά το θέμα της ασφάλειας είναι το ίδιο. Όλα τα πυρηνικά απόβλητα πρέπει να υπάγονται στους ίδιους κανόνες ασφαλείας. Έχουν δίκιο οι συνάδελφοι ότι οι οικονομικές πτυχές της διαχείρισης ε, ε, των αποβλήτων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Για τις μεγάλες αυτές γενικές γραμμές μπορούμε ίσως να κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις, αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η αρχή του ορυπαίνου πληρώνει. Εκείνος που είναι υπεύθυνο θα πρέπει να αναλάβει τα απόβλητα αυτά και θα πρέπει να κρατήσουμε στα χέρια μας τον έλεγχο όλης της αλυσίδας από τη μεταφορά μέχρι την τελική αναπόθεση. Και τέλος, Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, υποβάλαμε μία σειρά τροπολογιών και καμιά φορά η μετάφραση, η γραπτή αυτών των ε, τροπολογιών είναι κάπως περίεργη. Γιατί όταν θέλουμε να καταλήξουμε σε τελικές ε, συμβαστικές τροπολογίες πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην προσωρινή εναπόθεση και την τελική εναπόθεση και καμιά φορά η γραπτή μετάφραση του κειμένου δεν το δίνει αυτό. Επίσης κύριε Βιτάλ δεν συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι στις οδηγίες υπάρχει κάτι το πολυγενικό. Ε, όχι είναι σε θέση μια οδηγία να διακανονίσει κάποιους τομείς. Μπορούμε να στείλουμε κατά αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα προς όλα τα κράτη-μέλη. Οι εισηγήτρια νομίζω και οι ισιώδεις εισηγητές έχουν πολλά να κάνουν στις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κάθλιν, λέει ο πρόεδρε. Η Τζούντιτ Μέρκη είναι επόμενη στον κατάλογο και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Γκέρεκ που είναι ο το χειρότερο μέρο τη μέλος τη επιτροπή, να με αντικαταστήσει εδώ στο θόκο του Πρόεδρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να συμφωνήσω με την ε, συνάδελφο. Θα ήθελα να προσθέσω και κάποια άλλα πράγματα όμως. Ε, αν κοιτάξουμε τη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι κάθε κράτος μέλος ε, θα πρέπει να ασχολείται το ίδιο με την αποθήκευση ε, των πυρηνικών αποβλήτων, ενώ υπόθηκε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Αρκετοί συνάδελφοι το είπαν αυτό Ε, και αν κοιτάξουμε την ιστορία της Ευρώπης βλέπουμε ότι και η τα σύνορά μας ε, αλλάζουν. Αν κοιτάξουμε τις εξελίξεις των τελευταίων ε, 2.000 ετών, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η διάσταση των αποβλήτων δεν μπορεί να είναι εθνικό ζήτημα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, διαχείρισης των αποβλήτων. Ε, δεν λέω ότι μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα τις εθνικές αρμοδιότητες στο θέμα αυτό. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να ε, αντιμετωπίσουμε το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν κοιτάξουμε την αποθήκευση, εμένα στη χώρα μου υπάρχει πολύ λάσπη και πυλός. Εάν θέλουμε να χτίσουμε σπίτια, πρέπει να στηρίξουμε καλά τα θεμέλια στη Φιλανδία. Μπορεί κανείς να αποθηκεύσει ε, τα απόβλητα σε βάθος 3-4 ε, χιλιάδων ε, μέτρων, αλλά αυτό στη χώρα μου δεν γίνεται. Έχω λοιπόν πολλές παρατηρήσεις για το θέμα της υπόγειας αποθήκευσης ή διάθεσης, διότι θα πρέπει να σφραγίζονται ε, οι αποθήκες αυτές. Ε, δεν ε, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να μετακινηθούμε προς την υπόγεια αποθήκευση μέχρι να έχουμε μια οριστική λύση και δεν νομίζω ότι η λύση αυτή για την οποία μιλάμε είναι οριστική. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις συνθήκες, διότι αλλάζουν τα σύνορα, αλλάζουν οι γεωλογικοί σχηματισμοί, αλλάζει και το κλίμα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι δυνατόν να υιοθετήσουμε διάφορα μέτρα, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Δεν υπάρχει οριστική ασφάλεια ή ίστατη ασφάλεια όταν μιλάμε για υπόγεια αποθήκευση. Εάν δεν είναι ασφαλής, ε, λοιπόν, δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Δεν λέω ότι η επίγεια αποθήκευση είναι ασφαλής, ε, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να παρέμβουμε σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της επικοινωνίας, ε, διότι είδαμε τις ε, αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χίλια χρόνια. Μπορεί σε χίλια χρόνια από τώρα ο κόσμος να μην μιλάει την ίδια γλώσσα, πόσο μάλλον σε εκατό 100.000 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα της τελικής διάθεσης, θα πρέπει να μπορούμε και ε, να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους και στο μέλλον. Ε, αν λοιπόν εξετάσουμε την εθνική ασφάλεια θα πρέπει να γίνει γρήγορη η επικοινωνία αν ε, σχεδιάζουμε έναν χώρο τελικής εναπόθεσης διότι μπορεί κάποιοι τέτοιοι χώροι να επηρεάζουν και άλλα κρατημέλη. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει επικοινωνία. Επίσης, όταν μιλάμε για η υπόγεια αποθήκευση θα πρέπει να έχουμε σωστή επικοινωνία και θα πρέπει να παρακολουθούμε και την ε, υπόγεια ε, εναπόθεση, διότι αν μιλάμε για προσωρινή υπόγεια αποθήκευση και πάλι θα ήθελα να γνωρίζω περισσότερα για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Μέρκης. Κυρία Ριμπάς. Μικρόφωνο, παρακαλούμε. Voilà, sorry. Oui, je voudrais... Εισαγωγικά, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο όρους ε, που χρησιμοποιείτε. Μιλάτε για το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων και το θέμα της επεξεργασίας. Εγώ ήμουν βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Γαλλίας και έκανα μία ε, έκθεση για το θέμα της διαχείρισης ε, των πυρηνικών αποβλήτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επεξεργασία, μιλάμε για το φαινόμενο της μετάλλαξης και εδώ ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί με τη μετάλλαξη ε, δεν θα μπορούμε να τη διαχειριστούμε όλα. Πρέπει λοιπόν να μιλάμε για, θέμα, για διαχείριση ζεστιών, γιατί δεν μπορούμε να μειώσουμε τα απόβλητα. Το δεύτερο που μας απομένει στη διαχείριση των αποβλήτων είναι η αρχική παρέμβαση, ε, είναι η αναπόθεση ή η υπόγεια αποθήκευση. Δεν έχουμε ε, άλλες λύσεις. Και αυτά που θέλω να σας πω εισαγωγικά είναι ότι πρακτικά δεν έχουμε ε, κλείσει οριστικά ε, τα πυρηνικά εργοστάσια και όταν θα ξεκινήσουμε θα έχουμε χιλιάδες τόνους πυρηνικά απόβλητα. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να ορίσουμε τι σημαίνει πυρηνικά απόβλητα και ο ορισμός τώρα που προτείνει η Κομισιόν δεν αρκεί. Γιατί, γιατί αφήνει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο στα κράτη-μέλη. Καταρχή δεν ε, ασχολείται με τα ε, απόβλητα από τα ε, ορυχεία. Στην Γαλλία έχουμε χιλιάδες τόνους που προέρχονται από ορυχεία ουρανίου και δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά. Έχουμε επίσης τα στρατιωτικά απόβλητα. Πώς θα ε, έχουμε μια οδηγία που αφήνει εκτός τα, τα απόβλητα τα στρατιωτικά. Θα πρέπει να ενταχθούν στο θέμα της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων. Και υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο επί το οποίο δεν επιμένουμε και μιλάμε για το κατόφλι εξαίρεσης, ε, δηλαδή το κατόφλι κάτω από το οποίο δεν θα μιλάμε πλέον για πυρηνικό απόβλητο και πάνω από το οποίο θα έχουμε πυρηνικό απόβλητο. Εμείς είχαμε αυτό το πρόβλημα με ε, τις... Ε, με τις ράγες που ήταν ε, μολυσμένες. Αν δηλαδή δεν φτάσουμε ε, Παραδείγματο χάρη στο να καθορίσουμε ένα τέτοιο όριο ε, θα έχουμε πρόβλημα γιατί τι έκαναν ε, όσοι εκμεταλλευόταν είχαν ε, θέσει ένα όριο και είχαν ε, πει ότι δεν είναι πυρηνικά απόβλητα αυτά έτσι λοιπόν εκείνα τα υλικά τα διαχειρίζονταν ως κανονικά οικιακά απόβλητα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εδώ. Άλλο στοιχείο τη συζήτηση είναι η εξαγωγή των πυρηνικών αποβλήτων. Μας λένε και μίλησε κάποιος συνάδελφος ε, και είπε ότι αυτό δεν ανήκει στην οδηγία. Βεβαίω και είναι τμήμα τη οδηγία και μάλιστα στο άρθρο 4 ε, και πόσο μάλιστα που ο Επίτροπος ε, Έτιγκερ και αυτό είναι μήνυμα στην Κομισιόν ήταν σαφής και είπε δεν θα έχουμε εξαγωγέ προ τι τρίτες χώρε. Δεν θα έχουμε εξαγωγέ προ τι τρίτε χώρε. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χώρα θα πρέπει να διαχειρίζεται τα δικά της πυρηνικά απόβλητα. Και όταν αναφερόμαστε στην οδηγία του 2006, η οδηγία αυτή έχει ξεπεραστεί σήμερα γιατί τοποθετήθηκε ο Επίτροπος και είπε όχι εξαγωγές. Στη Γαλλία υπάρχει ένας νόμος για τα πυρηνικά απόβλητα που λέει δεν έχουμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε ξένα απόβλητα. Και ξέρετε ότι για χρόνια απόβλητα που έρχονται από Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο κτλ έφταναν ε, στο ΛΑΚ, στο πυρηνικό σταθμό εκεί και αποδοκεύονταν εκεί και θα έπρεπε τελικά ε, να καταβούν στα χαρακόμματα οι βουλευτές για να επανέλθουν στη χώρα τους ε, τα πυρηνικά απόβλητα. Έτσι λοιπόν εγώ συμφωνώ εδώ με τον Επίτροπο Έτιγκερ να μην έχουμε καμία εξαγωγή των αποβλήτων. Κάτι για το κόστος τώρα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα το κόστος των αποβλήτων. Ε, να ξέρετε ότι στη Γαλλία όταν ε, ε, αξιολογήσαμε το κόστος της υπόγειας αναποδεύσης μιλήσανε για 50 εκατομμύρια ευρώ και μετά από τρία χρόνια μίλησαν για 35 εκατομμύρια ακόμη δεν έχει κατασκευαστεί θα πρέπει λοιπόν ε, να είναι οι επιχειρηματίες που θέτουν χρήματα γιατί εμείς ε, να πληρώσουμε οι φορολογούμενοι και γιατί οι επιχειρηματίες ε, δεν θέλουν να κλείσουν τα εργοστάσια γιατί είναι τεράστιο το κόστος και θα πρέπει να είναι αυτοί όμως που θα το αναλάβουν οι επιχειρηματίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα περιμένουν, δεν θα τα κλείσουν τα εργοστάσια ή κάποια στιγμή θα τα κλείσουν και θα σου πούν «Α, να συνεισφέρετε κι εσείς». Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κάτι ακόμα ε, για τις ε, πισίνες. Ε, υπάρχουν κοντά στα πυρηνικά εργοστάρια τέτοιες πισίνες απόθεσης των αποβλήτων στη Γαλλία. Ε, λέμε παραδείγματο χάρη αργότερα θα γίνει η επεξεργασία. Όμως, τι μα έμαθε η Φουκουσίμα, όλοι αυτές οι χώροι απόθεσης δεν προστατεύονται με κάποιους ε, όρους ασφαλείας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια λοιπόν. Αν υπάρξει τρομοκρατική επίθεση, σκεφτείτε και έτσι παίρνουμε το σχάρι, για πέντε χρόνια αποθηκεύονται σε αυτά τα σημεία, γιατί πριν τα πέντε χρόνια δεν μπορούμε να τα πάρουμε ως πυρηνικά απόβλητα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα αν είμαστε υπερήκατα των πυρηνικών. Πρέπει να σκεφτούμε τις επόμενες γενιές. Έτσι λοιπόν ο, καλύτερος θα, ο καθένας θα πρέπει να διαχειριστεί στο δυνατόν καλύτερα αυτά τα απόβλητα ε, και να ορίσει τα απόβλητα αυτά. Ευχαριστώ κύριο Φάντσο. Ευχαριστώ. Λέω κύριο Σέντσου. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω με τη σειρά μου την άποψή μου. Συμφωνώ με όσους μίλησαν προηγμένως Ούτε εμεί ε, πρέπει να ξοδεύουμε ιδιαίτερη ενέργεια μιλώντας ε, για το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα εδώ συζητούμε ένα διαφορετικό θέμα και νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στον έλεγχο, στον πιο αυστηρό έλεγχο σε ό,τι αφορά στη διαχείριση αυτών των πυρηνικών αποβλήτων θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στον έλεγχο των μέτρων ασφαλείας σε σχέση με την αποθήκευση, με την αναπόθεση των αποβλήτων και ταυτόχρονα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των κρατών μελών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να βρεθούν νέες λύσεις σε ό,τι αφορά την αποθήκευση και τη μεταφορά των πυρηνικών αποβλήτων. Πιστεύω ότι καταρχήν θα πρέπει να ενισχύσουμε και την επιστημονική έρευνα σε αυτό τον τομέα για να εξεύρουμε νέες τεχνολογικές λύσεις με καλύτερες επιδόσεις και πιο ασφαλείς. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να προσδιορίσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια το επίπεδο ευθύνης όσων μεταφέρουν τα απόβλητα, όσων παράγουν τα απόβλητα, όσων τα αποθηκεύουν. Έχουμε αρκετά παραδείγματα, αρκετές περιπτώσεις ε, όπου τα κριτήρια και οι ισχύοντες κανόνες δεν έχουν γίνει σεβαστοί μέχρι τέλους. Και τα αποτελέσματα δεν ήταν στο ύψος των προσδοκιών μας. Και κάθε φορά κανείς δεν αναλάμβανε την ευθύνη. Πιστεύω ότι τα πρότυπα ασφαλείας, οι κανόνες ασφαλείας πρέπει να γίνονται σεβαστοί και πρέπει να προβλέψουμε πολύ ισχυρά μέτρα κατά όσων δεν σέβονται αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Και είναι αλήθεια ότι ε, τελικά με το φόβο μόνο ε, έχουμε αποτελέσματα, έτσι λέμε στη Ρουμανία, ίσως ε, και εδώ ταιριάζει αυτή η παροιμία, όμως εγώ νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν μιλάμε μόνο ε, για τη μεταφορά των αποβλήτων, αλλά μιλάμε και για τα πυρηνικά καύσιμα μεταξύ των κρατών μελών. Και αυτό ενέχει κίνδυνο. Και για να αλλάξω θέμα θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στη συνάδελφο κυρία Χέρτσοκ. Είναι σήμερα τα γενεθλιά τη. Ευχαριστώ πολύ. Και για την τελική σας δήλωση, την τελευταία σας δήλωση. Θα παρακαλούσα τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να ε, παρέμβει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια για την έκθεση. Νομίζω ότι σήμερα γίνεται μία εις συζήτηση για τα βασικά θέματα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα δεν ε, πιεζόμαστε από το χρόνο. Η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση σχετικά με την ε, διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Είτε είναι κανείς υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας, ε, θα πρέπει να γίνει η διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων. Το πρόβλημα αυτό βρίσκεται στην πόρτα μας και θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Ακόμα και αν σταματήσουμε την ε, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ε, με πυρηνική ενέργεια. Ε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας, διότι δεν θα φύγει από μόνο του το πρόβλημα. Αυτά είναι η ε, και ακούσαμε κάποια επιχειρήματα για την Φουκουσίμα. Εάν θα μπορούσα εγώ να βγάλω ένα συμπέρασμα και κάποιες παρεμβάσεις το έθιξαν αυτό, η Φουκουσίμα μας έδειξε τι μπορεί να γίνει με τα αναλωμένα καύσιμα που βρίσκονται σε δεξαμενές. Ε, πρέπει να γίνει η διαχείριση αυτών. Και ακριβώς το να αρνηθούμε την ε, οδηγία είναι αντιπαραγωγικό. Νομίζω ότι η νομική γνωμοδότηση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου είναι σαφής. Ε, λέει ότι ε, η συνθήκη Euratom καλύπτει το θέμα αυτό. σε αφορά τη, τους χρηματικούς πόρους, πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε και αυτό που προτείνει η Κομισιόν είναι... να υπάρχουν επαρκείς ε, πόροι όταν είναι απαραίτητοι για την ε, διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και διενεργών αποβλήτων, όπως ε, για παράδειγμα για την ε, δημιουργία ενός χώρου τελικής εναπόθεσης των αποβλήτων. Μπορούμε να επιβάλλουμε κάποιους περιορισμούς σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτών των χώρων, αλλά η οδηγία καθορίζει τους στόχους που πρέπει να πετύχουν τα κράτη-μέλη και στόχος είναι η οικονομική πόρη να είναι πρώτον επαρκής και δεύτερον να είναι διαθέσιμη εγκαίρως ώστε να λυθεί το θέμα που θα αντιμετωπίζουμε. Εάν το Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει ακόμα πιο πέρα, αυτό μπορεί να γίνει δεν ε, θα προσθέσει τίποτα όμως στους βασικούς στόχους που έχουμε. Άκουσα πολλές παρεμβάσεις ε, σχετικά με τους όρους ε, και τους ορισμούς. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες για το άρθρο 3 όπου έχουμε τους ορισμούς. Προσωπική μου έκκληση θα ήταν παρακαλώ κοιτάξτε πρώτα εάν είναι απαραίτητοι όλοι αυτοί οι ορισμοί. Εγώ είδα ότι προτείνονται κάποιοι όροι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται καν μέσα στην οδηγία. Παρακαλώ λοιπόν εξετάστε εάν οι όροι όντως είναι απαραίτητοι και ορισμοί και δεύτερον παρακαλώ προσπαθήστε να ευθυγραμμιστείτε με τους συμφωνημένους όρους που έχουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο διεθνές πλαίσιο. Εσείς προτείνετε να αλλάξει το γλωσσάριο της ε, Διεθνούς ε, Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας. Ξέρετε ότι από τεχνικής πλευράς ε, αυτό μπορεί να γίνει, διότι οι ορισμοί αυτοί ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη οδηγία. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να υπάρχει γενική συνέπεια στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Και στην, στο ευρύτερο πλαίσιο η διάθεση θεωρείται ότι είναι μόνιμη, ενώ η αποθήκευση προσωρινή. Ακούσαμε πολλές ε, παρεμβάσεις ε, σχετικά με τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Φυσικά, φυσικό είναι ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζομένους. Υπάρχουν όμως ήδη πολλοί τρόποι προστασίας των εργαζομένων. Και ο ειδικό τρόπος ε, είναι η ειδική οδηγία και το άρθρο 31 της συνθήκης Euratom που προβλέπει οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από την ε, ιονίζουσα ακτινοβολία. Επίσης, ανοίγει η πόρτα για την περιφερειακή συνεργασία. Αυτό ε, μπορεί να είναι χρήσιμο οικονομικά, γεωλογικά και όσον αφορά τη γενική πολιτική. Αλλά ένα πράγμα θα είναι απόλυτα σαφές. Όταν μιλάμε για περιφερειακή συνεργασία και συνεργασία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μιλάμε για εξαγωγή των αποβλήτων. Όσο παραμένουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μιλάμε για εξαγωγή. Και τίθεται το θέμα που όσο θέλετε να υπαγορεύετε συγκεκριμένα πράγματα στα πλαίσια αυτά. Η Κομισιόν με την πρότασή της επιτρέπει πολλή ευελιξία στα κράτη-μέλη για να πετύχουν το στόχο της περιφερειακής ε, διάθεσης. Μήπως είναι ε, αντιπαραγωγικό το να είμαστε υπερβολικά συγκεκριμένοι όσον αφορά αυτά που υπαγορεύουμε για την επίτευξη των ε, στόχων που θέλουμε να πετύχουμε. Και όσον αφορά την εξαγωγή ε, ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι αυτό που βλέπουμε εδώ δεν είναι μόνο μια πρόταση του κυρίου Τινέρη, είναι πρόταση του συνόλου του σώματος της Επιτροπής και Το σύνολο της Επιτροπής θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να εξάγονται επικίνδυνα απόβλητα. Έχουμε ήδη ε, νομοθεσία για την ε, απαγόρευση τοξικών αποβλήτων ε, μη πυρηνικών, αλλά τα πυρηνικά απόβλητα είναι τουλάχιστον εξίσου επικίνδυνα με τα άλλα τοξικά απόβλητα των οποίων απαγορεύεται η εξαγωγή. Ο Επίτροπος έχει καταστήσει σαφές ότι αν το Κοινοβούλιο θέλει να έχει τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και συμφωνεί με αυτό, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σε τρίτες χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία επιρροή στον τρόπο αποθήκευσης και διάθεσης των αποβλήτων. Και τέθηκε το ερώτημα προς ποιες χώρες ε, θα μπορούμε να εξάγουμε τα πυρηνικά απόβλητα και νομίζω ότι είναι σαφές. Εάν ζητήσουμε χώρους τελικής αναπόθεσης ε, για την διάθεση των αποβλήτων. Η απάντησή μου είναι ότι εγώ δεν γνωρίζω καμία χώρα όπου να υπάρχει ήδη χώρος τελικής εναπόθεσης ή που να λειτουργεί χώρος τελικής εναπόθεσης. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ζητήσει τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας όσον αφορά τα πυρηνικά απόβλητα. Η υψηλότερη ασφάλεια όμως δεν σημαίνει ασφάλεια 100%. Στον βιομηχανοποιημένο κόσμο στον οποίο ζούμε, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση 100%. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να συζητάμε το μείγμα ενέργειας, ε, τον ε, συνδυασμό πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούμε, διότι βρίσκεται εκτός ε, του εδώ στο πεδίο εφαρμογή ε, τη πρόταση που έχουμε μπροστά μα. Ε, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να έθιξα τα βασικά θέματα. που αναφέρονται στις τροπολογίες και ελπίζω μαζί με την κυρία Χέρτσο να καταλήξετε τόσο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια γνωμοδότηση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ και την Κομισιόν που μας έδωσε ξεκαθαρές απαντήσεις. Υπάρχει κάτι με το οποίο όλοι συμφωνούμε. Τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας δεν σημαίνουν 100% ασφάλεια και ελπίζω να αποσυρθούν όλες αυτές ε, οι τροπολογίες γιατί θα περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός τροπολογιών. Θα πρέπει να ψηφίσουμε άλλωστε επί τροπολογιών και τελικά θα είναι πιο ρεαλιστικό το κείμενο. Ήδη τόνισα ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στα πολιτικά κριτήρια. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γνώση και τις δεξιότητες που έχουμε ως πολιτικοί και θα πρέπει να αφήσουμε στους εμπειρογνώμονες να ρυθμίσουν όσα είναι υπό τη δική τους αρμοδιότητα. Νομίζω ότι δεν είναι κατάλληλο να λέμε ότι είναι κακή η οδηγία μας γιατί δεν αναφέρει τους λόγω ε, του σεισμού στη Φουκουσίμα ή λόγω του τσουνάμι. Νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς εννοούμε με αυτό, αλλά δεν πρέπει να κινηθούμε προς ε, ένα τεχνικό ορισμό όπου θα αναφέρουμε τις συγκεκριμένες απειλές. Ε, αυτός είναι ένας συγκεκριμένος τομέας που συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερα από σεισμούς και τσουνάμι. Μπορούμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά φαινόμενα που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και αν εισαγάγουμε μία ανάλυση για πιθανές τεχνικές λύσεις, τότε θα αποδυναμώσουμε την οδηγία. Συμφωνώ με την κυρία Χέρτσοκ συγκεκριμένα ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε εδώ, η προσθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι. Επίσης, ξέρω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τι είναι ρεαλιστικό, τι μπορεί να επιτευχθεί και τι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Πρέπει να παραδεχτώ ότι είμαι πιο φιλόδοξη εδώ από την Κομισιόν. Συμφωνώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι έχουμε επαρκή χρηματοδοτικά μέσα και είναι στη διάθεσή μας όταν χρειάζονται. Αλλά νομίζω ότι σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την αρχή ο πληρώνει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ή θα πρέπει να πετήσουμε ε, αυτοί οι χρηματοδοτικη πόροι να ενεργοποιούνται και να προσανατολίζονται προς το στόχο και πρέπει να έχουμε τους καταλλήλους ελέγχους, γιατί αν ε, δεν υπάρχει έλεγχος, πολλά μπορούμε να λέμε στην οδηγία, αλλά το θέμα είναι αν τελικά θα έχουμε εφαρμογή τη. Σε ό,τι αφορά τους ανεξαρτήτους εμπειρογνώμονες, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητος έλεγχος, Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ε, ρυθμιστικές αρχές, αλλά φυσικά ένας ορισμός πρέπει να βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια και όχι σε τεχνικά. Υπάρχουν πολλά άλλα ακόμα θέματα τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω, αλλά αν το πράξω αυτό θα επαναλάβω πράγματα που υπόθηκαν. Δεν θα το κάνω λοιπόν. Θα ήθελα να δω το Κοινοβουλίο να διαδραματίζει ένα μεγαλύτερο ρόλο από όσο διαδραμάτιζε μέχρι σήμερα. Αυτό αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους. Και φυσικά αυτό ισχύει και για την οδηγία αλλά και για τους ελέγχους. Όλοι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη Συνδική Ευρατόμ, η οποία μας ε, δίνει ορισμένες ε, προτεραιότητες και ορισμένα όρια. Ελπίζω το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη τη δική μας εργασία. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον κύριο Κούμπλιγκερ και ελπίζουμε ότι θα λάβουν το έργο μας υπόψη γιατί γνωρίζω ότι παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το χρονοδιάγραμμά μας έχει προσαρμοστεί. Έτσι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την κατάλληλη χρονική στιγμή Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε ε, να συντομεύσουμε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία γιατί πρέπει να έχουμε και μια επικοδομητική συζήτηση. Ελπίζω ότι στις 26 Μαΐου θα συζητήσουμε στην Επιτροπή αυτή το συγκεκριμένο θέμα και στις 23 Ιουνίου θα ψηφίσουμε στην ε, μήνυ Ολομέλεια εδώ στις Βρυξέλλες. Ελπίζω ότι αυτή αυτό το χρονοδιάγραμμα βρίσκεται σύμφωνο και το Συμβούλιο και ελπίζω και μάλλον πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα καταλήξει σε απόφαση αφού ψηφίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ε, εξαντλητική η συζήτηση, ελπίζω. Να σας υπενθυμίσω και πάλι ότι στις 26 Μαΐου θα ψηφιστεί το κείμενο στην Επιτροπή. Εδώ ολοκληρώσαμε το σημείο 3 της ημερησίας διάταξης και ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα να υποδεχτώ την κυρία Λεπερούς, να την καλέσω εδώ στο βήμα. présentation. <clears throat> Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη έχει να κάνει με την ε, έκθεση ομάδας εμπειρογνωμόνων που αξιολόγησαν την εφαρμογή του προγράμματος Eurostars. Να σας θυμίσω ότι το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε το 2008 και σχετίζεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Η γενική ιδέα είναι να φέρουμε την επιστήμη πιο κοντά στον οικονομικό τομέα. Η κυρία Λαπερούς είναι επικεφαλής της ομάδας επιρογνωμόνων. που έκανε την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος. Ε, σας καλωσορίζουμε και πάλι. Η κυρία Λαπερούς είναι πρώην συνάδελφός μας από την προηγούμενη θητεία. και ελπίζω να έχετε να μας παρουσιάσετε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή των ε, αποφάσεών μας. Είναι σπάνιο οι αποφάσεις ε, και τα ψηφίσματά μας να οδηγούν σε τέτοιου τύπου δράσεις. Και είναι σπάνιο να μπορούμε να ελέγξουμε αν είχαμε δίκιο όταν λαμβάναμε τις αποφάσεις αυτές. Δίνω το λόγο λοιπόν στην κυρία Λαφερούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είδα πολλού που γνωρίζω και άτομα με το οποίο έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Είναι πραγματική ικανοποίησή μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου έκανε τη μήνα με διορίσει πρόεδρο αυτή τη ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματο Eurostars. Θα σας ε, το παρουσιάσω. Πόση ε, χρόνο έχω στη διάθεσή μου, ένα τέταρτο, θα, με πείτε, θα μου πείτε αν ε, μακρηγορήσω. Έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο έθεσε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα Eurostar τον Ιούλιο του 2008, από τον Ιούλιο του 2008 στο 2013 και σύμφωνα με την απόφαση αυτή θα πρέπει να γίνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν το πλαίσιο και ε, την οργάνωση και τις κυρίες συστάσεις, ε, αλλά θα αναφερθώ και στην ε, υλοποίηση του προγράμματος. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από τον Ιούλιο ως τον Νοέμβριο του 2010 και η τελική έκθεση υπευλήθη το Δεκέμβριο του 2010 και δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Απριλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έκανε και συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Εδώ βλέπετε την ε, ομάδα των εξάρτητων εμπειρογνώμων. Ε, ο κύριος Ερκο Ότιο είναι ο εισηγητής, είναι καθηγητής και επίσης έχουμε και την Μάγια Μπουγκάρ που είναι συνεισηγήτρια και συνέταξε μέρο τη έκθεση. Ε, στη συνέχεια, Γιώργ Λίκτ ε, είναι πανεπιστημιακό, ακαδημαϊκό, ε, που έχει ειδικεύσει στι μικρέ και μισέ επιχειρήσει. Ο κ. Χωσέ Μολέρο έρχεται από την Ισπανία. Επίση, είναι καθηγητή, συμμετέχει ιδιαίτερα στην έρευνα για τι μικρέ και μισέ επιχειρήσει. Και η κυρία Λένα Τσπούρη είναι επίση καθηγήτρια από την Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή αξιόλογου εμπειρογνώμονε για την υλοποίηση αυτή τη αξιολόγηση. Αυτά είναι τα κυρία θέματα τώρα στα οποία έπρεπε να απαντήσουμε για να αξιολογήσουμε τη θέση εφαρμογή του προγράμματος Eurostars. Η πρόοδος, ε, η πρόοδος που έγινε σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος, ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, ε, ε, η πρόσβαση των μικροκομιστών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα αυτό και Ποιε ήταν επιδόσεις αυτού του προγράμματος σε ό,τι αφορά ε, την ένταξή του στα εθνικά προγράμματα, αξιολογήθηκε προς το αξία του προγράμματος και κατόπιν ε, αξιολογήσαμε τη σημερινή πολιτική και υλοποίησαμε συστάσεις για την περίοδο 2011-2013 και συστάσεις για μετά το 2013 και φυσικά ε, αξιολόγηση μέτρηση του γενικού αντίκτυπου του προγράμματος. Δηλαδή αν ε, αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών, ε, αν αυξήθηκε ο ρυθμός ε, των διπλωμάτων βρυστεχνίας που κατατέθηκαν κτλ. Σε αυτά να αναφερθώ σε λίγο. Εδώ στη συνέχεια αναφέρω την περιγραφή του προγράμματος. Έχει να κάνει με την έρευνα και την ανάπτυξη στις ΜΜΕ σε ό,τι αφορά τις νέες διαδικασίες, νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα τα σχέδια που κατατέθονται πρέπει να έχουν τεθεί στην αγορά μέσα σε τρία χρόνια, να είναι προσανατολισμένα στην αγορά δηλαδή. Υπάρχουν ε, ελάχιστοι συμμετέχοντες, δύο χώρες, ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, δύο ε, χώρες εταίροι. Σήμερα έχουμε 32 χώρες στην ομάδα και ο κύριος συμμετέχοντας ε, πρέπει να είναι μία ΜΜΕ που αφιερώνει τουλάχιστον 10% του κύκλου εργασιών στην έρευνα και στην ανάπτυξη και το πρόγραμμα το διαχειρίζεται η γραμματεία της πλατφόρμας Εύρικα. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100 εκατομμύρια ευρώ και η συμμετοχή των κρατών είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για όλη την περίοδο. Ε, μία μικρή μέση επιχείρηση είναι ένας εταίρος ε, μιας επιχείρησης ε, που θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα, συστήνεται συνήθως να έρθει σε επαφή με τον εθνικό συντονιστή NPC, National Project Coordinator λέγεται στα αγγλικά και στη συνέχεια θα υποβάλει την ε, πρόταση ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Γιουρίκα, του Εύρικα. Υπάρχει μια κεντρική αξιολόγηση που υλοποιείται καταρχήν από τεχνικούς εμπειρογνώμονες και στη συνέχεια από ένα ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων που καταρτίζει ένα κατάλογο κατάταξης ανάλογα με το επίπεδο ποιότητας ε, των project και κατόπιν έχουμε τις τελικές διαπραγματεύσεις ε, για τη σύμβαση που υλοποιείται με το Εθνικό Φορέα Χρηματοδότησης. Πρόκειται για τον οργανισμό που χρηματοδοτεί και παρακολουθεί το project αυτό. Κάποια αριθμητικά στοιχεία, πρόκειται για στοιχεία από το Δεκέμβριο του 2010 που μας έδωσε η γραμματεία του Γιουρίκα Έχουμε 1127 ε, προγράμματα που λάβαμε για ε, τις η ε, προσκλήση υποβολής προτάσεων που είχαμε, έχουμε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ένα χρόνο, έχουμε 1566 εκατομμύρια ευρώ και 3.790 συμμετέχοντες. Το ποσοστό ε, των ΜΜΕ που αφορούσαν ήταν το 72%. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας από τους στόχους εδώ έχει επιτευχθεί. Είχαμε 458 σχέδια που επιλέχθηκαν, ήταν πάνω από το κατόφλι ποιότητας, ε, καθώς αυτά συνήθως χρηματοδοτούνται και αυτό αφορά 329 project που εγκρίθηκαν για τη χρηματοδότηση και το Δεκέμβριο είχαμε και 14 προγράμματα που ολοκληρώθηκαν. Μιλάμε, αν σκεφτείτε ότι μιλάμε από το 2008, χρειάστηκε κάποιος χρόνος. Ε, είχαμε χρηματοδότηση από το κράτη-μέλη 85 εκατομμύρια ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 28,6 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα 6 εκατομμύρια ευρώ ε, δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους εθνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης. Εδώ έχουμε τα κύρια μηνύματα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινοτομία, γιατί είδαμε ότι το 70% των συμμετεχόντων είναι ΜΜΕ. Πετύχαμε το στόχο λοιπόν. Σε επίπεδο επιτυχίας το 25% των προτάσεων που υποβάλλονται επιλέγονται για τη χρηματοδότηση και ε, μιλάμε για νέα προϊόντα, νέες διαδικασίες και υπηρεσίες που είναι κοντά στην αγορά. Αυτό επιτρέπει μια εξέλιξη των ε, προώθησης των τεχνολογιών και του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο και ε, είδαμε ότι το σύστημα διακυβέρνησης ήταν πολύ καλό και μάλιστα βελτιώθηκε και από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα αυτό. Στη συνέχεια μας είπαν μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Είχαμε πολλές συνεντεύξεις με τη γραμματεία του Γιουρίκα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, με τις ενδιαφερόμενες ΜΜΕ. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μας επέτρεψαν ε, να ε, καταλήξουμε σε αυτά τα αποτελέσματα σήμερα. Τα πανεπιστήμια και επιχειρήσεις μας είπαν ότι η πρόσβαση ήταν πάρα πολύ εύκολη η αξιολόγηση που υλοποιήθηκε σε κεντρικό επίπεδο είναι πολύτιμη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την εκτιμούν αντίθετη διαδικασία για τη χρηματοδότηση γιατί ε, οι συμμετέχοντες πρέπει να απευθυνθούν στο εθνικό σημείο επαφής είναι κάπως πιο δύσκολη γιατί υπήρξαν κάποιες αποκλήσεις ε, στις διάφορες οργανώσεις, στους διάφορους οργανισμούς μεταξύ των χωρών. Είχαμε χώρες που ήταν ήδη πολύ οργανωμένες, ενώ άλλες που έπρεπε να συστήσουν ε, τις διαδικασίες για τη χρηματοδότηση. Είχαμε λοιπόν κάποιες χώρες όπου υπήρχαν μεγαλύτερες δυσκολίες. Τα εθνικά σημεία επαφής ε, και ο εθνικός συντονιστής του προγράμματος είναι πολύ σημαντικά για τους συμμετέχοντες γιατί ουσιαστικά στην, βοηθούν στην υλοποίηση, ε, δηλαδή και για τη χρηματοδότηση, για την απόκτηση της χρηματοδότησης ή για την υπογραφή της σύμβασης με τον εταίρο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που είναι από κάτω προς τα πάνω. Σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν υπάρχουν ε, θεματικές, μπορούν να εξεταστούν όλα τα θέματα. Είναι πολύ ευρύ ως προς την εφαρμογή λοιπόν και δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Αυτές είναι οι βελτιώσεις που προτείνουμε μέσω της αναλυσής μας. Ε, τώρα, εξιολόγηση που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι η βάση εμπειρογνωμόνων, ε, των τεχνικών εμπειρογνωμόνων πρέπει να εμπλουτιστεί. Σήμερα η γραμματεία του Γιουρίκα το Ευρικά που διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα διαθέτει ε, από 500 700 τεχνικούς εμπειρογνώμονες ε, και ε, αυτό ε, μας φαίνεται ότι μπορεί να είναι επαρκές σε ό,τι αφορά τις, ότι μπορεί να μην είναι επαρκές σε ό,τι αφορά τις γνώσεις οικονομικό και κοινωνικό τομέα και θεωρούσαμε ότι ίσως θα μπορούσε να υπάρχει και ένα σύνδεσμος με ένα άλλο πρόγραμμα και η ανάλυση που γίνεται από το πάνελ των εξάρτητων των εμπειρογνωμόνων θα έπρεπε να μας επιτρέψει να υπάρχει περισσότερος χρόνος για την ανάλυση των διάφορων ε, προγραμμάτων. Αυτό μας είπε μάλιστα ο πρόεδρος ε, του πάνελ των εξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Επίσης, οι συμμετέχοντες ε, θα ήθελαν να έχουν περισσότερο feedback για την τεχνική αξιολόγηση, έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλουν ένα πρόγραμμα και αν ε, δεν έχουν επιλεχθεί ε, να μπορούν ε, να βελτιώσουν την πρότασή τους για την επόμενη φορά. Επίσης, σε εθνικό επίπεδο πρέπει να γίνει πρόοδος. Ορισμένα κράτη ο απαραίτητο χρόνος μέχρι την υπογραφή της τελικής συμφωνίας, της τελικής σύμβασης χρηματοδότησης, πολλές φορές ε, είναι αρκετά μεγάλη η χρονική περίοδος αυτής και μπορεί να καθυστερήσει το project. Επίσης είναι σημαντικό ε, να υπάρχει feedback ε, και ενημέρωση μεταξύ των σημείων επαφής και της γραμματείας του Γιουρίκα, του Ευρικά. Και στη συνολική αξιολόγηση αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε ότι τα project που επιλέχθηκαν τελικά πάνω από το επίπεδο ποιότητας ε, φτάνουν στο 63% ως το 80% για τις χρηματοδότησεις. Ελπίζουμε ότι ε, αν χρηματοδοτούμε ε, προϊόντα πάνω από ένα επίπεδο θέλουμε όλα να χρηματοδοτούνται. Εδώ έχουμε από 63% 80%. Επίσης έχουμε το θέμα του time to contract, δηλαδή από τη στιγμή που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ο φάκελος στη γραμματεία του Γιουρίκα μέχρι να ξέρουμε ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση, ότι θα χρηματοδοτηθεί και να γίνουν συμφωνίες των κοινοπραξιών. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλο αυτό το χρονικό διάστημα, ανάλογα με τα κράτη και είναι κάπως κρίμα γιατί εμείς ενθαρρύνουμε project που πρέπει να έχουν τεθεί στην αγορά μέσα στα τρία έτη. Τι διαπιστώσαμε από πολλούς επιλεχθέντες συμμετέχοντες ήδη έχουν μία εμπειρία σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς ε, προσπαθήσαμε ε, να έχουμε μια μεγαλύτερη γκάμα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, αξιολογήσαμε τις επιδόσεις ε, για την ένταξη στα εθνικά προγράμματα. Ξεκολουθούν να παραμένουν διμερεί συμφωνίες που δεν έχουν υπογραφεί μεταξύ γραμματείας Γιουρίκα και των εθνικών χρηματοδοτικών φορέων. Υπάρχει το πολύ σημαντικό θέμα που το αποκαλούμε το εικονικό κοινό ταμείο. Αν χρειάζεται ένα πραγματικό ή ένα εικονικό τέτοιο ταμείο, common pot, ε, τώρα τα κράτη δεσμεύονται σε ένα επίπεδο συγκεκριμένο επίπεδο προπολογισμού και περιμένουν πρακτικά οι επιχειρήσεις του ίδιου τους του κράτους ε, να λάβουν το ίδιο το ποσό να το ανακτήσουν. Έχουμε, αν είχαμε ένα κοινό ταμείο, δεν θα είχαμε παρετήτως την επιστροφή των χρημάτων που έχουν δοθεί. Σήμερα έχουμε κατά κάποιο τρόπο ένα εικονικό κοινό ταμείο, τελικά δηλαδή χρηματοδοτούν τα κράτη ακριβώς ε, με το ποσό του προϋπολογισμού που έχουν ανακοινώσει στις επιχειρήσεις τους ή στα πανεπιστημία τους, στους συμμετέχοντες του κράτους τους. Επίσης, είδαμε ότι ήταν απαραίτητο να εναρμονίσουμε καλύτερα τους κανόνες χρηματοδότησης. Ε, το ποσοστό χρηματοδότησης είναι λιγότερο σημαντικό. Μπορεί να έχουμε κράτη που χρηματοδοτούν ως το 40% αλλά ως 75% δεν ε, υπάρχει κάτι στάνταρ εδώ, αλλά αυτό δεν με συνοχλεί. αλλά οι κανόνες χρηματοδότησης, ναι, αν αποφασίσουμε να χρηματοδοτήσουμε πανεπιστήμια με θα έπρεπε σε όλα τα κράτη να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Κατόπιν είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε και τις χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται σε επίπεδο, τα κονδύλια που χορηγούνται σε επίπεδο κράτους και το κάναμε αυτό σε επίπεδο γραμματείας. Σήμερα μετά τα δύο έτη εξακολουθούν να τρέχουν τα προγράμματα και η, τα κονδύλια, η χρηματοδότηση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, υπάρχει, δεν έχουν ακόμη δοθεί. Υπάρχει δηλαδή μια χρονική απόκληση. Οι εμπειρογνώμονες μας είχαν μια δυσκολία να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Από όσα, μας, από σας είπα, διαπιστώνουμε ότι ήταν επιτυχές το πρόγραμμα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό για να έχουμε ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες και να ενθερρύνουμε ακόμη περισσότερο την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα σας προβληματίσει και στα πλαίσια του 8ου προγράμματος πλαίσιο τώρα κόστος όφελος αυτού του προγράμματος ε, σήμερα. Έχουμε το 6% του κόστους της διαχείρισης μας φαίνεται λογικό. Φυσικά όσο περισσότερους συμμετέχοντες, περισσότερους συμμετέχοντες έχουμε, μάλλον θα αυξηθεί και τα κόστος. Μίλησα για το κοινοταμείο, τώρα ορισμός του time to contract χρόνος μέχρι την υπογραφή της σύμβαση. Είναι πιο τεχνικό το θέμα αυτό. Το συζητήσαμε με τη Γραμματεία και με την Κομισιόν για να δούμε πώς ορίζεται. Εμεί μιλάμε για το χρόνο που τρέχει από τη στιγμή που υποβάλλει την πρόταση από την επιχείρηση και μέχρι τη στιγμή ε, της σύναψης της σύμβασης. Επίσης, ε, παρακολούθηση των δαπανών ανάλογα με το καθεστώς ε, του προγράμματος και αυτό πρέπει να παρακολουθείτε ε, από την Γραμματεία και από την Κομισιόν έτσι ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει και να αποζημιώσει η Κομισιόν τα κράτη που έχουν δώσει τα κονδύλια κατόπιν πρόθεση και μάρκετινγκ του προγράμματο. Το ίδιο και εδώ. Ξέρουμε ότι ήταν επιτυχέ το πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι η τάση είναι να έχουμε όλο και περισσότερου συμμετέχοντε, αλλά όσο περισσότερη πρόθεση έχουμε για να φτάσουμε και σε τέρους που δεν έχουν ευρωπαϊκή διεθνή εμπειρία, τόσο περισσότερο θα χρειαζόμαστε χρηματοδότηση. Είναι μια επιλογή που πρέπει να γίνει λοιπόν και ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γραμματεία. Για μα είναι ξεκάθαρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα και, το... και αναθέτει την εκτελεσή του στη Γραμματεία του Γιουρίκα. Σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων πιστεύουμε ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν επιτυχές ε, στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, θα πρέπει να συνεχιστεί. Ανάγκη εναρμόνισης και στήριξης ε, σε εθνικό επίπεδο. Επίσης ε, ζητούμε να υπάρχουν περισσότερα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή για να γίνεται καλύτερη αξιολόγηση του προγράμματος ε, γιατί ε, τώρα είμαστε στη μέση, μόνο 14 προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί, δεν μπορούσαμε λοιπόν να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο για τον αριθμό των προγραμμάτων που έχουν κατατεθεί και για τον αριθμό θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί. Οι ΜΜΕ μας είπαν ότι ήταν ικανοποιημένες αλλά δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτή την την αξιολόγηση. Μας φαίνεται λοιπόν σημαντικό και αυτό να τεθεί σε εφαρμογή από τη γραμματεία του Γιουρίκα, του Εύρικα και επίσης εναρμόνιση των εθνικών κανόνων και των κανόνων χρηματοδότηση είναι απαραίτητη. Αυτά μπορώ να σας πω σήμερα. Συμπερασματικά, συστάσεις. Πρέπει να υπάρχουν επαρκή κονδύλια για να έχουμε ίσως περισσότερα προγράμματα που να χρηματοδοτούνται πάνω από το επίπεδο ποιότητας, γιατί είπαμε ότι χρηματοδοτούνταν ε, από το 60% στο 80% των προγραμμάτων άνω του κατοφλίου ποιότητας. Ε, ίσως θα μπορούσαν να συνεισφέρουν και τα κράτη-μέλη με προς το προπολογισμό, ίσως θα μπορούσε να το συζητήσει αυτό και η Κομισιόν και στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου, γιατί εν μέρει χρηματοδοτείται αυτό από το πρόγραμμα συνεργασίας. Κατόπιν ε, η που δεν έχουν ακόμη ε, διεθνή εμπειρία, να φροντίσουμε να μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να αυξηθεί ο αριθμός των τεχνικών εμπειρογνωμόνων, ε, να υπάρχει ε, παρκές feedback στους συμμετέχοντες και να μειωθεί ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, γιατί μιλάμε για προϊόντα που τίθεται στην αγορά, να εναρμονιστούν εθνικοί κανόνες, και επίσης να ρυθμιστεί το θέμα του εικονικού κοινού ταμείου, του Common Pot. Εμείς προτείναμε σήμερα το 10% ε, του εικονικού ταμείου να τεθεί σε ένα πραγματικό κοινό ταμείο για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν περισσότερα project άνω του κατοφλίου ποιότητας και αν δεν δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια ε, να χορηγηθούν στη συνέχεια σε μια κατοπινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων και να τεθούν σε εφαρμογή τα μέτρα για να αξιολογηθεί καλύτερα ο αντίκτυπος. Ήμουν πολύ ικανοποιημένη που εργάστηκα σε αυτό το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαθεσιμότητά της, ε, την ε, εμπειρογνωμοσύνη, την αυστηρότητα. Εκτίμησα πάρα πολύ αυτή την αυστηρότητα και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και τη γραμματεία του Γιουρίκα Είχαμε πολύ πλούσιη ανταλλαγή απόψεων και μπορώ να πω ότι θα γίνουν, ε, θα σημειωθεί περαιτέρω αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι για τα δύο χρόνια είδαμε ότι πολύ γρήγορα τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα και η Ευρώπη μπορεί να είναι αποτελεσματική για τις ΜΜΕ και θα πρέπει να εργαστείτε ακόμη περισσότερο για τις μικρές και ευαισθητές επιχειρήσεις και να τους συμπεριλάβετε αυτό στον προβληματισμό σας για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Λαπερούζο για την πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική αυτή παρουσίαση. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Η κυρία Χέρτσοκ πρώτη έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί ξέρουμε, τι θα έρθουμε να ακούσουμε την κυρία Περούς όταν ξέρουμε ότι ό,τι κάνει δεν το λαμβάνει κανένας από εκεί πάρει υπόψη του. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Η δική μας επιτροπή πάντα είναι υπέρ των γνώσεων, υπέρ των ΜΜΕ. Γι' αυτό το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους και επειδή μελλοντικά θα συζητήσουμε το ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο για την έρευνα και την κεντρονομία είναι νομίζω η σωστή χρονική στιγμή αυτή να έχουμε όλα τα επιχειρήματα στα χέρια μας ότι θα πρέπει να γίνει και τι, ε, θα μπορούμε να, πώς θα μπορούμε να συμβάλλουμε για να είμαστε πιο επιτυχείς. Έχω ορισμένες ερωτήσεις. Συμφωνώ ότι η χρηματοδότηση και οι διάφορες μέθοδοι της χρηματοδότησης στα κράτη-μέλη μπορούν να οδηγήσουν στρεβλώσεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω Πώς συγκρίνεται αυτή την ενδεχόμενη στρέβλωση με την ε, συνεπή εξέλιξη αναπεριφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα νέα κράτη-μέλη, υπάρχουν επικρίσεις για τα ε, θεσμικά όργανα, αλλά εάν οι στρεβλώσεις οφείλονται στην τοπική χρηματοδότηση, δεν ξέρω πώς ε, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Δεύτερον, θα με διέφερε να ξέρω σε ποιους τομείς υπάρχουν οι επιτυχίες. Ποιοι είναι οι κύριοι συμμετέχοντες. Μπορούμε να το πούμε ή είναι διασπαρμένα και λίγο πολύ παντού. Τρίτη ερώτηση. Αυτές οι εταιρείες που συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό πώς συμμετέχουν σε πληροφορίες για άλλα σχέδια. Πώς μπορούν δηλαδή να φτάσουν να χρησιμοποιούν περισσότερους πόρους ε, ή μπορούν να είναι Ξέρω ότι κάτι μας είπατε, αλλά μπορείτε να μας το εξηγήσετε καλύτερα και ω εισηγήτρια για την ε, νομική πράξη για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτά που έχετε κάνει μέχρι στιγμή και για την προετοιμασία για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Dziękuję bardzo. Ε, Pan de Campos. Κύριος Κάμπος έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι που είχα άλλε ενηλυμένες υποχρεώσει ε, και έχασα ένα τμήμα τη παρουσίαση, ε, Πρέπει να πω ότι μου αρέσει πολύ το πρόγραμμα ευρικά όταν ε, τώρα εμείς όλοι αφαισιωνόμαστε και, θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία μέσω των ΜΜΕ, βρισκόμαστε ενώπιον ε, μιας τυπικής ε, κατάστασης όπως του Μελέρου, ο οποίος ε, ουσιαστικά έκανε ένα διάλειμμα και με τη διαφορά όμως ότι όσοι έκαναν την πρόζα ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Έτσι λοιπόν, ε, το πρώτο μήνυμα είναι να δηλώσω πόσο ικανοποιημένο είμαι από την αξιολόγηση αυτή. Είναι πολύ λεπτομερής και πολύ αντικειμενική και θα θέλαμε ε, επίσης ε, να γίνεται το ίδιο και με άλλα προγράμματα. Όμως η ερώτηση που θέτω είναι το εξή. Εμείς τώρα εδώ λαμβάνουμε πολιτικές αποφάσεις για την επιστήμη και για την καινοτομία για το πρόγραμμα πλαίσιο 8. Και Έχουμε εδώ μία περίπτωση ποιότητας και μπορώ να πω και μία ιστορία επιτυχίας. Τώρα η ερώτηση που θέτω είναι εξή. Πώς αυτή η ιστορία επιτυχίας ε, δεν διευρύνεται ε, και ε, τι θα γίνει στο μέλλον με το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Δηλαδή έχουμε ακριβώς το ίδιο σύστημα ε, πόρων θα δώσουμε στο Εύρυκα αυτή τη χρηματοδότηση σε αυτές τις 32 χώρες ε, και όλα λειτουργούν πολύ καλά, δεν χρειάζεται να ενσυχούμε οι αξιολογήσεις πάντοτε είναι πολύ καλές, όλα τρέχουν πολύ καλά, όλα βαίνουν ομαλά. Όταν δεν υπάρχουν ειδήσει είναι καλά τα νέα. Αλλά παρόλα αυτά, μήπως εδώ χάνουμε μια ευκαιρία για να αναπτύξουμε και να διευρύνουμε περισσότερο ε, αυτό το πρόγραμμα. Περισσότερο στην Κομισιόν απευθύνουμε, όχι σε εσά. Ελπίζω και η Κομισιόν να έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να παρέμβει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να υποβάλω μια ερώτηση. Ε, θα ήθελα κάπως να εμβαθύνω το θέμα, το οποίο έφτιαξε η κυρία Χέρτσοκ. Θα ήθελα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τους 14 αυτούς προσανατολισμούς στους οποίους αναφερθήκατε όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται άμεσα με την αγορά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, τον κύριο Ράχιαρτ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν καλωσορίζει την έκθεση από την εξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, τις οποίες ε, προεδρεύει η κυρία Λαπερούζ. Συγχαιρόμαστε την ομάδα αυτή για την εργασία της. δεν ήταν πάντα εύκολο να, πετύχουν, να πετευθούν στόχοι και συνεπή στοιχεία. Ε, πρέπει να είστε σίγουροι ότι η Κομισιόν θα ε, εξακολουθήσει να υποστηρίζει το πρόγραμμα αυτό μέχρι το 2013 όπως προβλέπετε από τον κανονισμό και όπως προβλέπετε και στον ε, οικονομικό φάκελο. Δεν θέλω να κατασπατελίσω το χρόνο σας. Η κυρία Λαπερούζ αναφέρθηκε που χρειάζονται περισσότερες βελτιώσεις. Οι ΜΜΕ που έχουν διεθνή εμπειρία είχαμε ήδη μια απάντηση. Δηλαδή αντί από εδώ να περνάνε οι επιχειρήσεις σε, άλλες, σε άλλα προγράμματα, μάλλον το αντίθετο γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν εδώ κάτι να διορθωθεί ίσως. Επίσης υπάρχουν πολλά προγράμματα που θα πρέπει να ενδυναμωθούν. Τα στοιχεία ενημέρωσης ε, δίνονται στην έκθεση αξιολόγησης και το θέμα του τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον εξαρτάται από τις συζητήσεις που γίνονται όχι μόνο μέσα στα πλαίσια του πολιτού ε, δημοσιονομικού πλαισίου αλλά και στις συζητήσεις για τη μελλοντική το μελλοντικό στρατηγικό πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια δημόσια αξιολόγηση που τελειώνει τέλη Μαΐου. Και μετά στην Κομισιόν θα αναλύσουμε τα μέσα που θα υπάρχουν, θα συνεχιστούν δηλαδή οι συζητήσεις και στο ιστορικό της Επιτροπής και μεταξύ Επιτροπής και του σώματος εδώ για να υποστηριχθούν καλύτερα οι ΜΜΕ. Αν νομίζω ότι η κοινή συμφωνία υπάρχει, ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται έντονη ενίσχυση. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε την υποστήριξη για τις ΜΜΕ στα μελλοντικά προγράμματα Πράγμα που δεν είναι αυτονόητο γιατί υπάρχουν και άλλα συμφέροντα. Και δεν πρέπει να ξεχάμε ότι οι ΜΜΕ είναι εκείνε που καθορίζουν την οικονομική ταυτότητα της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Λαπερούς και να την παρακαλέσω να απαντήσει στις ερωτήσει που υπευλήθησαν και να μας παρουσιάσει σχετικές τις απόψεις. Λοιπόν, όσον αφορά την ερώτηση Edit, για τους κανόνες χρηματοδότησης, δεν ξέρω αν είχατε την περιέργεια να μελετήσετε το παράτημα 10 της έκθεσης που αναφέρει του, τους κανόνες ανά έτος, ανακράτο συγγνώμη, είναι διαθάσιμη εκεί. Επίσης, οι κανόνες στην ιστοσελίδα του Eurostars. Υπάρχουν εκεί διαφανώς όλοι οι κανόνες. Τυχαία εγώ παίρνω τώρα, χωρίς να κάνω αξιολόγηση, Αυστρία. Η Αυστρία χρηματοδοτεί μέχρι 60% της ΜΜΕ 60% μπορεί να είναι μικρές, 40% μέσο μεγέθους, τα πανεπιστήμια μπορούν να φτάσουν μέχρι το 60%, οργανισμοί ερευνά 80%. Να μεταβλέπω βλέπω εδώ. Την Ουγγαρία, Φερρυπίν. ΜΜΕ μέχρι 25%, πιο μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι 5% και τα πανεπιστήμια μέχρι 100%. Μετά τι να πάμε, τη Γαλλία, που δεν χρηματοδοτεί τις μεγάλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, κάθε φορά η κατάσταση είναι διαφορετική. Παραδείγματο χάρη, ο Γάλλο εταίρο δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί με έναν Έλληνα εταίρο, γιατί οι κανόνε τη Ελλάδα δεν είναι ανάλογοι με του κανόνε που υπάρχουν στη Γαλλία που παραδείγματος χάρη δεν χρηματοδοτείται το πανεπιστήμιο. Λυπηρό αυτό κάπως. Οι διαφορές δεν είναι γεωγραφικού τύπου, είναι οι διαφορές λόγω των κανόνων χρηματοδότησης. Η Ελβετία, παραδείγματος χάρη, δεν χρηματοδοτούσε τη ΜΜΕ. Ανάγκαστηκε λοιπόν να προσαρμόσει το σύνταγμά τη για να μπορέσει να τη χρηματοδοτήσει. Αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για εναρμόνιση των κανόνων οι τομείς όπου υπάρχει η μεγαλύτερη επιτυχία, στο πίνακα 3 της έκθεσης αναφέρατε αυτό ανατομέα. 19 νέα στις θαλάσσιες μεταφορές, 23 αγροτική βιομηχανία τροφίμων, 450 εφαρμογής ε, τεχνολογία πληροφορικής, και 73 ε, στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Και μπορώ να κάνω και προσωπικά δύο παρατηρήσεις. Βιοτεχνολογία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαδικασία είναι πολύ πιο μακροχρόνια, ενώ για τις ε, τεχνολογίες ε, πληροφορικής η επιτυχία είναι πολύ πιο γλυγορή, 6 μήνες περίπου παραδείγματο χάρη μια επιχείρηση με την οποία ήρθα, σε επαφή είπε ότι αν δεν είχε χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωστάρ δεν θα μπορούσε να προσλάβει 30 μηχανικούς. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον τομέα τους ε, βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τους Ινδούς και τους Κινέζους. Εάν δεν μπορούσε να έχει προσλάβει τους, 30 δηλαδή θα είχε διακυβευτεί και κινδυνεύσει όλη η επιχείρηση. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να υπάρχει αξιοπιστία έναντι των τραπεζών, παραδείγματος χάρη για τις επιχειρήσεις αυτές. Επίσης έχουν ένα σήμα ευρωπαϊκό αν θέλετε, για να μπορέσουν να περάσουν σε διαδικασίες τις οποίες καμιά φορά δεν θα μπορούσαν να έχουν μπει. Αυτή η επιχειρήση στην οποία αναφέρομαι ήταν κάπως στα σύνορα της ε, χρηματοδότηση γιατί από τον ε, κύκλο εργασιών τους αυτό το σχέδιο ήταν το 25% περίπου, δηλαδή θα μπορούσε δεν θα μπορούσε να το χρηματοδοτήσει από μόνη της. Λοιπόν, αυτοί που κερδίζουν είναι πολύ ευχαριστημένοι. Βέβαια, μπορεί κανένας να αναρωτηθεί αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Σέντρα παραδείγματο χάρη ήταν ήδη ένα πρόγραμμα πλαίσιο για να ενθαρρυνθούν οι ΜΜΕ, να ενταχθούν. Λοιπόν, οι ΜΜΕ είτε στο πρόγραμμα συνεργασία είτε στα θεματικά προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν. Ε, καμιά φορά λένε ότι ναι, αλλά εμεί θέλουμε να συμμετάσχουμε κάπως ε, μας συνθλίβει ένα πρόγραμμα πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που ανταποκρίνει στις δικές μας δυνατότητες. Γι' αυτό είναι καλύτερο εδώ να έχουμε ένα πρόγραμμα στα δικά μας μέτρα, αν θέλετε. Κάπως έτσι σχηματικά σας το παρουσιάζω, αλλά νομίζω ότι η εικόνα είναι σωστή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε εκτός αυτού ότι μία ΜΜΕ έχει σαν ρόλο να κερδίσει χρήματα. Πρόκειται για business. Πολύ περισσότερο βέβαια παρά αν στρεφόμαστε προς τις πανεπιστήμια ή και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν μακρά εμπειρία ανάπτυξης και έρευνας. Οι ΜΜΕ θέλουν αμέσως αποτελέσματα βέβαια. Κάνουν έρευνα και ανάπτυξη, και αυτό σχηματικά σας το λέω, αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και μετά το θέμα των πόρων, το είπατε δικαίως. Και η Κομισιόν το είπε. Σήμερα όλοι με την οικονομική κρίση που δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα, κοιτάνε τα πράγματα πολύ προσεκτικά. Ξέρουμε ότι μπορούν πολλά χρήματα να, να χρησιμοποιηθούν ή να χρηματοδοθεί η έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πού. Ε, για το πρόγραμμα πλαίσιο άκουσα τη σύσταση των εμπρογνωμών που είναι τουλάχιστον να διατηρηθεί ο προπολογισμό. Δεν ξέρω πώς θα τύχει διαχείριση λοιπά. Ορισμένες χώρες μας είπαν ότι προτίθεται να αυξήσουν το ποσοστό τους. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αυξήσει, ίσως ορισμένα κράτη-μέλη να αυξήσουν. Θα το κάνουν τουλάχιστον για το τρέχον πρόγραμμα. Γιατί οι δεσμεύσει του προπολογισμού θα ξεπεράσουν αυτό που υπήρχε μέχρι στιγμής, από ό,τι είδαμε εφαρμογές σχετικά με την αγορά είχα ακριβώς κατά νου αυτή την επιτυχή ε, ιστορία. Εκείνο που μας είπαν ότι όχι μόνο μπορέσαμε να βρούμε πελάτες, μας επέτρεψε επίσης η χρηματοδότηση. Οι εταίροι μας να γίνουν πελάτες μας κατά κάποιο τρόπο. Αυτά. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λαπερούζ. Νομίζω ότι ε, ένα είναι το σαφές συμπέρασμα της έκθεσης αυτής. Ε, το πρόγραμμα αυτό πληρεί τους στόχους του. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, θα γίνουν κάποιες προσαρμογές, ε, φαίνεται όμως ότι θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Όσον αφορά την συνέχεια του, Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε στο επόμενο στάδιο του προγράμματος αυτού, όπου θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε τα επιτεύγματα του προγράμματος αυτού σε δύο χρόνια από τώρα. Κύρια Λαπερού, σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας, για την εκθεσή σας και να σας ευχηθώ. Ε, δημιουργικό έργο και στο μέλλον. τη δουλειά σα ε, πάνω στα ζητήματα αυτά τα οποία είναι τόσο σημαντικά για την αγορά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, σχεδόν τελειώσαμε τη σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε φτάσει στα διάφορα. Δεν είναι εδώ ο πρόεδρος της Επιτροπής μας σήμερα. Δεν έχουμε κανένα θέμα στα διάφορα. Να σας θυμίσω απλά ότι την επόμενη εβδομάδα θα συμμετάσχουμε σε πολύ σημαντική συνεδρίαση της Επιτροπής μας που θα ε, συμπεριλαμβάνει ψηφοφορίες. 9 Μαΐου λοιπόν έχουμε ψηφοφορίες στο Στρασβούργο. Και τέλος, Νομίζω ότι το μόνο που απομένει είναι να σας ευχαριστήσω όλους ε, και να πω ότι λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.